ψηφοφορίες θα ήθελα να προαναγγείλω κάτι. Ο κύριος Σέντεγκάτ γνωστοποίησε ότι από τις 5 Φεβρουαρίου 2014 <clears throat> καταθέτει την εντολή ως Ευρωβουλευτής. Το Ευρωκοινοβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 4 εδάφιο 3 του κανονισμού του διαπιστώνει την χειρία της έδρας από, την 5η Φεβρουαρίου 2014 και το Κοινοβούλιο ενημερώνει σχετικά και την αρμόδια Εθνική Αρχή περί τούτου. Κυρίες και κύριοι, τώρα θα ξεκινήσουμε με τις ψηφοφορίες. Στην ημερήσια διάταξη έχουμε την έκθεση του κυρίου Μορέιρα.